Έχουν έρθει και δύο για να ανταλλάξουμε απόψεις ε, για ε, τα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ της δημοκρατίας και, της, ε, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκονζάτο που βρίσκεται εδώ σήμερα, που είναι πάντα στην διάθεσή μας και που πάντα με τόση όρεξη συνεργάζεται με την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να σας παρουσιάσω την κοινή ανακοίνωση η οποία τονίζει την πρόταση του είπα του Αντιπροσώπου και της Κομισιόν για ένα νέο σχέδιο δράσης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας παρουσιάσω το πλαίσιο. Το σχέδιο δράσης αυτό στόχο έχει να αντικαταστήσει το σχέδιο δράσης ε, που εξέπνευσε στο τέλος του 2014 και αποτελεί μέρος του πακέτου το οποίο προώθησε ιδιαίτερα το δικό σας κοινοβούλιο και το οποίο καθορίζει το στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία, το οποίο παραμένει ως έχει. Και επίσης έχει παραταθεί η εντολή του Σταύρου Λαμπρινίου, κάτι για το οποίο χαιρόμαστε ε, όλοι πάρα πολύ. Να σας πω πώς καταλήξαμε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Όταν έφτασα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ε, θέλησα να υπάρχει αίσθημα οικειοποίησης του σχεδίου δράσης αυτού. Και βέβαια ο βασικό ενδιαφερόμενο εδώ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό συνεργαστήκαμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα με την Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ για να εξολογήσουμε σε τι βαθμό ε, πετύχαμε τους στόχους που είχαμε θέσει. Προσπαθήσαμε να μάθουμε και κάποια πράγματα από το προηγούμενο σχέδιο δράσης. Ένα από τα πράγματα που μάθαμε ήταν ότι πρέπει να είναι πιο επικεντρωμένο, πιο στρατηγικό. Και η ανάγκη για πιο στρατηγικού στόχου οφείλεται στο γεγονό ότι θέλαμε ένα σχέδιο δράση το οποίο να αντιστοιχεί καλύτερα στην εντολή τη παρούσα Κομισιόν. Σημαντική είναι η ενδιάμεση αναθεώρηση, διότι θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε συντονισμό ανάμεσα στο σχέδιο δράσης και στα ε, χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα περάσουν από ενδιάμεση αναθεώρηση το 2017, διότι πολλοί από τους στόχους που θέτουμε δεν είναι μόνο πολιτικοί, ε, συνδέονται και με την χρηματοδότηση. Συνεπάγονται δηλαδή διοχέτευση της χρηματοδότησης προς τις σωστές κατευθύνσεις. Η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ λοιπόν έκανε τον ε, συντονισμό και με βάση την αξιολόγηση αυτή Θελήσαμε να καθορίσουμε τη νέα δομή και τους νέους στόχους. Αυτό λοιπόν έγινε σε συνεργασία με τις Γενικές διευθύνσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης προσπαθήσαμε στο βαθμό που είναι δυνατόν να πετύχουμε τη συμμετοχή και των άλλων ενδιαφερομένων. Παρουσίασα την προσέγγιση στο Κοινοβούλιο, στα κράτη-μέλη και στην κοινωνία των πολιτών είχα διάφορες συναντήσεις μαζί τους, όχι μόνο με την Τρόικα, αλλά με όλα τα μέλη του δικτύου. Ταυτόχρονα, πρέπει να σεβαστούμε την επιθυμία της Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι η πρωτοβολία παραμένει δική της και του είπα του αντιπροσώπου Γι' αυτό δημοσιεύσαμε πρώτα την πρόταση αυτή πριν την επίσημη διαβούλευση. Πού βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαβουλεύσεις με εσά, με τα κράτη-μέλη και θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις μας και με την κοινωνία των πολιτών με στόχο να υιοθετήσουμε αυτό το σχέδιο δράσης με συμπεράσματα του Συμβουλίου πριν το καλοκαίρι. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου σχεδίου δράσης. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω με την παρατήρηση ότι ε, αντιμετωπίζουμε όλο και πιο πολλές προκλήσεις στο περιβάλλον μας, κάτι το οποίο ε, ζούμε και στις διμερείς επαφές μας ε, και σε πολυμερή πλαίσια. Έχετε πάει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και παρότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα κατά την τελευταία σύνοδο, οι εταίροι μας μας παρουσιάζουν όλο και περισσότερες προκλήσεις. Τι προκλήσεις είναι αυτές. Καταρχάς, ε, αμφισβητείται η οικουμενικότητα των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, για πολιτιστικούς λόγους. Ακούμε όλο και περισσότερο ότι ναι, αλλά στη χώρα μας έχουμε άλλες παραδόσεις. Αμφισβητούνται και από το γεγονός ότι υπάρχουν νέοι διεθνείς παράγοντες που αμφισβητούν την πολυμερή προσέγγιση πιστεύουν ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να αποφαίνεται όσον αφορά την κατάσταση σε διάφορες χώρες. Υπάρχουν μη κρατικοί φορείς ε, με τους οποίους αρχίζει και γίνεται προβληματική η λογοδοσία για παράδειγμα. Ε, επίσης, στην κοινωνία των πολιτών ε, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Για παράδειγμα, συχνά χρησιμοποιείται η καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, ως δικαιολογία για περιορισμό του χώρου της ε, κοινωνίας των πολιτών. Και επίσης δείτε την κατάσταση στην ε, Μεσόγειο. Είναι μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και είναι ένα από τα θέματα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με το νέο σχέδιο δράσης. Με το νέο σχέδιο δράσης θέλουμε να συλλογιστούμε περισσότερο για το πώς μπορούμε να κάνουμε τις δράσεις μας πιο αποτελεσματικές. Θέλουμε δηλαδή να Έχουμε μια σειρά εργαλείων, μπορώ να σας αναφέρω τις κατευθυντήρες γραμμές, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τον διάλογό όμως για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε να φροντίσουμε να υπάρχει καλύτερη επαφή, καλύτερη ανταλλαγή ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα, μεταξύ άλλων και του διμερούς και του πολυμερούς. Έχουμε εντοπίσει λοιπόν τους πέντε τομείς δράσης που έχετε μπροστά σας. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι κατά τη γνώμη μου η προώθηση της οικειοποίησης από τοπικούς παράγοντες και με τις επαφές μου που έχω διαπιστώνω ότι και για πολλούς ε, είναι σημαντικό αυτό. Θα πρέπει από μέσα και όχι με εξωτερική πίεση να πείσουμε τους εταίρους μας να κάνουν περισσότερα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και γι' αυτό προσπαθούμε να εντατικοποιήσουμε τις επαφές μας και με κυβερνήσεις, με οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητους φορείς, δικαστικούς φορείς και μη κυβερνητικού οργανισμούς υπό το φως των αυξανόμενων απειλών που αντιμετωπίζει η κοινωνία των πολιτών σε πολλές χώρες. Ο δεύτερος τίτλος μάλλον θα είναι πιο προβληματικός διότι προσπαθούμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας ε, στις βασικές θεματικές προκλήσεις, τις οποίες θα πρέπει να τις δούμε σε σχέση με τους παράγοντες. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η ελευθερία λόγου είναι πάρα πολύ σημαντική, έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Την σχέση, για παράδειγμα, με την ελευθερία του συνεταιρίζεστε κλπ. Ε, έχουμε την καταπολέμηση των διακρίσεων, που επίσης λαμβάνει διαφορετικές μορφές, αλλά υπό τον τίτλο αυτό ε, σκεφτόμαστε ιδιαίτερα τις ε, γυναίκες, ε, τα άτομα ΛΟΑ, τα παιδιά και γενικά τις μειονότητες, όπως τις θρησκευτικέ μειονότητες. Και άλλο σημαντικό θέμα που νιώσαμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να προ, προβάλλουμε ε, ακούγοντας την κοινωνία των πολιτών ήταν η καταπολέμηση των βασανιστήριων υπό το φως των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι χώρες που είχαν εφαρμόσει το μορατόριουμ έχουμε επικεντρωθεί και στην ε, κατάργηση της αντικής ποινής μέσα στην επόμενη πενταετία. Επίσης, ε, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Η εμπειρία μας μας δείχνει ότι στους διαλόγους μας με χώρες εταίρους για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να βρούμε κάποια σημεία εισόδου και πιστεύουμε ότι τα κοινωνικά δικαιώματα είναι συνήθως καλύτερο σημείο εισόδου, μας επιτρέπει να έχουμε πραγματικό διάλογο και όχι απλά μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ κοφών. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δικαιώματα ως σημείο εισόδου και μετά να περάσουμε στα άλλα. Κατόπιν έχουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε περιπτώσεις συγκρούσεων και κρίσεων. Αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα. Είναι δύσκολο να βρούμε μία κατάλληλη ανταπόκριση, αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε το θέμα. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις κρίσεις γύρω μας. Θα πρέπει να ε, έχουμε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, ε, να έχουμε εργαλεία αποτροπής των κρίσεων και να επικεντρωθούν περισσότερο στα ανθρώπινα δικαιώματα στις ε, αποστολές μας στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ και θα υποβάλουμε και νέες προτάσεις υπό τον τίτλο αυτόν, είμαι βέβαιος. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι το κρίσιμο είναι αυτό που αντιμετωπίζει το πρόβλημα αξιοπιστία που αντιμετωπίζουμε. Έχει να κάνει με περισσότερη συνοχή και συνέπεια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί επανειλημμένα. Το εμπόριο είναι σημαντικό στοιχείο, όπως και η μετανάστευση. Είχαμε εντοπίσει τους τομείς αυτούς ε, πριν ε, την ακμή τη κρίση. Ε, Δυστυχώ η πραγματικότητα μας επιβεβαίωσε του φόβου μας και κατόπιν έχουμε την ε, αντιτρομοκρατία. Και ο πέμπτος ε, τομέα έχει να κάνει με τον πολιτισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία. Εδώ υπάρχουν διάφορες πτυχές. Έχω Ε, συμμετάσχει σε διάφορους ε, διαλόγους ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω ότι αυτοί οι διάλογοι θα πρέπει να ενσωματωθούν στα διάφορα κανάλια επικοινωνίας που έχουμε με τους εταίρους μας. Δεν θα πρέπει να είναι ξεχωριστή και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης των διμερών και πολυμερών πτυχών των εργασιών μας. Για παράδειγμα, στην Τίνιδα πριν λίγες μέρες μπορέσαμε να θίξουμε κάποια θέματα που συνδέονταν με την τελευταία σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρά τις ε, καλές σχέσεις μας με την, ε, την Ισία, είχαμε κάποιε διαφορές. Έτσι λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τις ε, θέσεις μας στην πρωτεύουσα και όχι μόνο στην Γενέβη. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη και Περιμένουμε τα κράτη-μέλη να υποβάλουν προτάσεις για δράσεις, ιδιαίτερα δράσεις υπό την δική τους ευθύνη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν περισσότερο ε, αίσθημα οικειοποίησης ε, και ε, και πρέσβεις μου έχουν εκφράσει τη θέση αυτή. Θα υποβάλουμε λοιπόν περισσότερες προτάσεις για το θέμα αυτό. Επίση, θα έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε ανησυχίε και του δικού σα κοινοβουλίου και τη κοινωνία των πολιτών. Προσλέπω στην καλή συζήτηση. Ζητώ συγγνώμη, θα πρέπει να αποχωρήσω στι 10 παρα 10. Είμαι όμω στη διάθεσή σα μέχρι τότε. όπω και ο Αντώνη, άλλωστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τι ερωτήσει μα, Η κυρία Λοκάμα έχει το λόγο πρώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτό το σχέδιο δράσης που είναι πολύ σφαιρικό, πολύ λεπτομερές πρέπει να σας πω πως δεν ήθελα να εστιάσω μόνο στα σημεία για το οποίο έχω επικρίσεις, αλλά και σε κάποια άλλα τα οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω. Πολύ σωστά εντοπίσατε τις περιοχές όπου χρειάζεται περισσότερη πολιτική στράτευση και που πρέπει να χαράξετε προτεραιότητες. Πάντως το σχέδιο δράση εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σφαιρικό. Χρειάστηκε να αφήσετε κάτι εκτός όπως είπατε και εσείς αντιμετωπίζετε πολλές προκλήσεις. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αν μπορείτε να μας πείτε να ξεκαθαρίσετε το εξής. Πώς αποφασίσατε το τι θα αποτελέσει προτεραιότητα. Στο σχέδιο δράσης έχετε συμπεριλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις των κρατών μελών. Γίνεται αυτή τη στιγμή συζήτηση κάπου Υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη επίσης έχουν την υποχρέωση αναφοράς για το πώς εφαρμόζουν τις διάφορες δράσεις ή σε ποιο βαθμό έχουν ε, ε, υλοποιήσει τις δεσμεύσεις τους, για παράδειγμα σε μια κοινή ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καινούριο βέβαια το θέμα, αλλά ίσως μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες προσπάθειες. Πολλέ δράσεις δεν συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Λέει συνεχιζόμενο, για παράδειγμα. Αυτό είναι ε, δίδαγμα του παρελθόντος. Γιατί ξέρετε πως αν δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, είναι πολύ πιο δύσκολο να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη για εμάς. Κάτι στο οποίο θα ήθελα επίσης να σταθώ μάλλον επικριτικά είναι πως το προηγούμενο σχέδιο δράσης είχατε πολλή στήριξη ε, για τη δημοκρατία στις ε, πιλωτικές χώρες, κάτι το οποίο μοιάζει να λείπει. Το θέμα αυτό το αναφέρεται στο σημείο 32, αλλά πουθενά αλλού, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την τοπική κυριότητα του προγράμματος, έτσι ώστε οι εθνικές ε, οργανώσεις που στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα να εμπλακούν πιο ενεργά. Οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ στην πολιτική, ε, στην εξωτερική πολιτική, στην πολιτική γειτονία ε, δίδουν ιδιαίτερη σημασία στο σημείο αυτό. Επίσης, τη δυνατότητα των κοινοβουλίων και των σωμάτων κατά της διαφθοράς στα κράτη αυτά. Είναι πολύ σωστό να έχουμε μια πολιτική που θα είναι ανοιχτή σε αυτούς τους θεσμούς. Κάτι που λείπει, κύριε Γκονζάτο, είναι το τι θα κάνουμε ε, για τα κοινωνικά οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Εκεί ίσως δεν το έχετε σκεφτεί επαρκώς. Μπορούμε να έχουμε πιο συγκεκριμένες δράσεις, για παράδειγμα, δικαίωμα σε καθαρό νερό, σε υπηρεσίες υγείας, Ένα επόμενο θέμα στο οποίο έχουμε σταθεί και στο παρελθόν είναι το δικαίωμα στην κυριότητα γης. Έχουμε κάποιους ε, που, ανθρώπους που υπερασπίζονται ανθρώπινα δικαιώματα και μόνο αυτοί έχουν συμπεριληφθεί στο σχετικό θέμα. Ε, θα έπρεπε λοιπόν κάπως να το ενισχύσουμε έτσι ώστε ε, το σημείο αυτό να φανεί περισσότερο. Ε, επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα νομίζω και εκεί χρειάζεται να μιλήσουμε περισσότερο για την εταιρική λογοδοσία. Πάντα υπάρχει μία πολύ δύσκολη διακριτική γραμμή που χωρίζει την εταιρική λογοδοσία από την ευθύνη, από την ατομική ευθύνη. Εκεί πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά. Επίσης, τι συμβαίνει με τις παραβιάσεις αυτού του, της νομοθεσίας από τις εταιρείε πώς μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για το μηχανισμό επιτήρησης αυτών, με ποιο τρόπο θα ε, τηρείται ενήμερο το Κοινοβούλιο. Γιατί στην προηγούμενη θητεία λάβαμε ελάχιστες πληροφορίες για το θέμα και νομίζω ότι μας εκπλήσει το ότι το συμπεριλαμβάνεται εδώ. Ε, λογοδοσία και μεταβατική δικαιοσύνη. Θα πρέπει ίσως να μιλήσουμε για τους στόχους μας, δηλαδή να μην υπάρχει ατιμορρησία για το σοβαρό ε, διεθνές έγκλημα και προστασία θυμάτων, αποζημίωση θυμάτων κτλ. Μήπως θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε το ποιοι είναι οι στόχοι μας εδώ. Στην παράγραφο 21α μιλάτε για δράσεις για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διεθνές ε, Δικαστήριο, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θα ήθελα να μου πείτε γιατί ενδιαφέρει και εμένα και τους υπόλοιπους συναδέλφους που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Παρακολουθούμε το τι συμβαίνει με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ίσως εδώ θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να γίνει μια δημόσια έκθεση αξιολόγησης με συγκεκριμένες συστάσεις έτσι ώστε να ε, συζητήσετε το θέμα με εμάς αλλά και με την κοινωνία των πολιτών. Στο τέλος της 21α μιλάτε για διευκόλυνση συμμετοχή, συνεργασία και πρόσβαση ε, των ενδιαφερομένων κρατών στο Διεθνές Ποινικό ε, Δικαστήριο. Νομίζω ότι αυτό γίνεται συχνά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ίδιο που κάνουμε για τα θέματα που αφορούν την θανατική ποινή. Οπότε γιατί γίνεται εδώ αυτή η ξεχωριστή αναφορά. Για το τελευταίο σχέδιο, το προηγούμενο σχέδιο δράσης, εκεί μιλήσατε για μία δέσμευση για τη μεταβατική δικαιοσύνη η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα ήθελα να μου πείτε πώς εξηγείτε την καθυστέρηση και αν υπάρχει κάποια εξήγηση. Θέλουμε και μία δέσμευτη ε, για να ε, έχουμε καθολική δικαιοδοσία ε, και στα εθνικά δικαστήρια κρατών αν έχουμε κάποια κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα έπρεπε να προβλέπετε και αυτό αφού έχουμε και τον ειδικό εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά, ίσως λοιπόν θα έπρεπε ο στόχος αυτός να συμπεριληφθεί στο σχέδιο δράσης για τις αποστολές ε, στο εξωτερικό. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Μήπως θα έπρεπε να αναφερθούμε και σε δυνατότητα ανακρίσεων, ερευνών και προστασίας καταδοτών. Επίσης, για τους πρόσφυγες είναι δύσκολο να το συζητήσουμε τώρα. Ας δούμε τι θα φέρει η μεγάλη συνδιάσκεψη στις 13 Μαΐου, γιατί σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτές οι προσεγγίσεις μου φαίνονται μάλλον περίεργες. Δηλαδή, το να μπορούμε να καταστρέφουμε σκάφη, ας πούμε, με ψήφισμα του ΟΗΕ, δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Τις εγκληματικές οργανώσεις θα πρέπει να τις καταπολεμήσουμε με άλλο τρόπο, αλλά αυτό καταλαβαίνω πως πρόκειται για μια πολιτική δήλωση από πλευρά μου. Ίσως και εδώ υπάρχει θέμα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη μετανάστευση να δούμε τι γίνεται και με τους συνοριοφύλακες και τη Frontex στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω και άλλες συστάσεις εδώ. Τι γίνεται με τους μετανάστες ε, στις χώρες από τις οποίες περνάνε πριν φτάσουν στην Ευρώπη. Και να μπούμε σε λεπτομέρειες. Γιατί δεν έχουν δυνατότητα καταγγελίας της Frontex οι πρόσφυγες ή οι μετανάστες αν θεωρούνται ότι κακοποιούνται για τους διακινητές και το τράφικινγκ. Εδώ θα λάβουμε μία έκθεση. Η στόχευση ακόμα αφορά τις χώρες προτεραιότητας. Ίσως όμως θα έπρεπε να δούμε γιατί κάποιες χώρες θεωρούνται χώρες προτεραιότητας. Στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική δεν έχω να κάνει κάτι με την πραγματικότητα εκείνης της χώρας παρά μόνο με το πόσο μετανάστες ε, έχει στη συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα, Τρίδες. για τα θέματα αυτά και για όσους δεν έχουν χαριά, χαρτιά όπως επίσης την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση μεταναστών από τρίτες χώρες, να σας πω πως η παρουσίαση ε, για το θέμα αυτό, για τα πάτριδας έχει συζητηθεί επαρκώς και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ε, συμπεριλάβουμε κάτι άλλο. Για την αντιτρομοκρατία, ε, για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, ίσως θα έπρεπε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση και για τα σημεία 27. Το σημείο 27 για την αξιολόγηση αντικτύπου και το πώς επηρεάζει τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου νομίζω πως το Μάρτιο η διαμεσολαβήτρια της Ευρώπης είπε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε την αναγκαία μελέτη αντικτύπου για την περίπτωση Βιετνάμ και πως αυτό αποτελεί παραβίαση. Καλό θα ήταν λοιπόν αυτές οι αξιολογήσεις να γίνονται. Βασανιστήρια. είπατε πως αποτελεί μία από τις θεματικές σας προκλήσεις. Στο σχέδιο δράσης θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Οι ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων επίσης δεν περιγράφονται με πολύ φιλόδοξη διατύπωση. Πείτε μου λοιπόν αν θέλετε να εφαρμόσετε την, ε, τις δεσμεύσεις για τα αναπτυξιακά κριτήρια και τέλος δεν έχουμε καμία καμία αναφορά για το τι γίνεται με τον αθλητισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χτες συζητήσαμε και με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και με το θέμα της ΦΥΒΑ. Μας είπαν, μα καλά, τι ακριβώς ρόλο έχουμε να παίξουμε εμείς. Ίσως δεν το κατανοούν ακόμα και θα πρέπει να τους εξηγηθεί. Ε, señora... Πεσέρα, θέλετε το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Γιατί η προλαλήσασα νομίζω δεν άφησε και πολλά για να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Και δεν ξέρω ούτως ή άλλως αν ο κύριος από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής θα μπορέσει να έχει χρόνο να απαντήσει. Θέλω να εστιάσω σε ένα στοιχείο το οποίο μου φαίνεται σημαντικό για το σχέδιό σας, που είναι η σημασία που δίνεται στην αξιοπιστία. Η μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη και την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση είναι η αξιοπιστία και μερικέ φορέ η δυνατότητα να την ανακτήσει εκεί που την έχει χάσει και να τη διατηρήσει εκεί που την έχει. Η αξιοπιστία στα ανθρώπινα δικαιώματα πετυχαίνεται μέσω, α, μέσα από έργα, από πράξεις και πρέπει να διατηρήσουμε την καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο, η βασική πρόκληση του σχεδίου. Μια πολύ, μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Και ποια είναι η απάντηση της Ένωσης έναντι προβλημάτων, πώς να τα πω, τραγωδίες, δράματα. Το, την τρομακτική πρόκληση της μετανάστευσης. Ποια είναι η απάντηση. Εκεί συγκλίνουν όλα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διπλωματίας. Υπάρχουν πολλά στοιχεία στο σχέδιό σας που φύγουν αυτό το θέμα. Θα ήθελα να μου πείτε όμως συγκεκριμένα ποια είναι τα σημεία επί των οποίων μπορούμε να εργαστούμε συνολικά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανθρώπινα δικαιώματα, ανάπτυξη, και εμείς και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, τέλος πάντων ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη κυρίως αυτό το δίπτυχο. Ο κ. Παντζέρη. Δεν είμαστε σε φάση τροποποίησης του σχεδίου. Θα ήθελα να καταλάβω κάποια πράγματα καταρχήν. Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω. Το, να, το πώς μπορούμε να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα, μια πολιτική φιλοσοφία αν θέλετε, ε, και κυρίω επί τριών πραγμάτων να στείλουμε αυτό το μήνυμα. Γιατί ούτως ή άλλως, για να το πω έτσι, αφήστε με να το πω έτσι, πρέπει να το πουλήσουμε και προ τα έξω αυτό το έγγραφο. Το θέμα δεν είναι να είμαστε σωστοί στο έγγραφο ε, σε σχέση με ό,τι έχει συμβεί. Το θέμα είναι να, να έχει και μια πρακτικότητα, έτσι. Καταρχάς, το θέμα της καθολικότητας τα πράγματα τα οποία γράφεται θα πρέπει να γίνουν βασικό στοιχείο της πράξης και της δράσης όλων των επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς, ας με γράφουμε αυτό, αύριο το πρωί θα συζητήσουμε για το TTIP και θα πάμε προς άλλη κατεύθυνση. Οπότε, τι νόημα έχει. Το δεύτερο στοιχείο είναι η λειτουργία η λειτουργία μας. Και για την πολιτική ατζέντα. Και για το, τη νέα πρόκληση που είναι η μετανάστευση, εμείς θέλουμε να ενισχυθούν οι αντιπροσωπείες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλες οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Η Φεντερίκα Μοντερίνη λέει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε, ας πούμε, την αντιπροσωπεία μας στον Ήγηρα. Πώς θα το κάνουμε. Έτσι. Θα πρέπει να προσδιορίσουμε αυτά τα πράγματα πάρα πολύ συγκεκριμένα. Η ενίσχυση λοιπόν των αντιπροσωπιών μας. Και τρίτο στοιχείο, το συζητήσαμε και χθε όταν μιλήσαμε για την Κεντρική Ασία. Θα πρέπει να βάλουμε νέα κριτήρια ερεσιμότητας. Γιατί τα παρελθόντα σε πολλές περιπτώσεις δεν λειτουργούν. Αν ήμασταν σε θέση να στείλουμε τρία πολιτικά μηνύματα και να, να δείξουμε ότι θα κάνουμε μια στροφή, γιατί βάζουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως βασικό στοιχείο της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοινοβουλίου, της, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, θα είναι καλά, καλό. Από εκεί και πέρα ας ε, τελειοποιήσουμε αν θέλετε αυτό το κείμενο. Το βασικό θέμα είναι να στείλουμε το μήνυμα πάνω απ' όλα όμως. Το... Η τελειοποίηση έρχεται μετά. Δεν ξέρω τώρα πώς θέλετε να απαντήσετε. Εσείς αποφασίζετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Συμφωνώ με αυτά που μόλις είπε ο Πιερ Αντώνιο Παντσέρη. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Το σχέδιο δράσης είναι ένας κατάλογος δράσεων και η δυσκολία είναι να είναι πολιτικά επίκαιρος αυτός ο κατάλογος. Το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης ε, θα υιοθετηθεί με συμπεράσματα του Συμβουλίου μας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλουμε ένα πολιτικό μήνυμα. Και με τα συμπεράσματα αυτά να τονίσουμε την φιλοσοφία στην οποία βασίζεται το νέο σχέδιο δράσης. Εκτιμώ τα στοιχεία που τονίσατε. Δεν ξέρω πώς να το πω στα αγγλικά. Ε, θα το πω στα ιταλικά. Η καθολικότητα. Θα πρέπει να εμπλακούν όλοι οι επίτροποι οριζόντια. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Σε αυτή τη φάση δοκιμάζουμε αυτή τη δομή μάλιστα. Και συμφωνώ επίσης ότι οι αντιπροσωπείες θα πρέπει να παίξουν ένα ρόλο. Οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να ενισχύσει την παρουσία της ε, και τη δυνατότητα που έχει να κάνει κάποια πράγματα στις διάφορες χώρες. Αλλά αυτό τι σημαίνει. Ε, πολύ στενή συνεργασία με την Κομισιόν, ε, γιατί όταν μιλάμε για θέματα μετανάστευσης δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, δεν είναι της υπηρεσίας εκτορικής δράσης, είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν. Και φυσικά θα πρέπει να συνεισφέρουν και τα κράτη-μέλη για να δοθούν απαντήσεις στο πρόβλημα της μετανάστευσης. Προς την Μπάρμπαρα Βελόχ Μπίλερ, πολλά από αυτά που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας. Δεν σας κρύβω ότι είχα και εγώ την ίδια την αίσθηση για τα οικονομικά και κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, ότι πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Ελπίζω όμως ότι σε αυτή τη φάση της διαδικασίας που είμαστε τώρα, όπου ερχόμαστε σε διαβούλευση με διάφορους ε, φορείς και με το Κοινοβούλιο, θα έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Και εκτιμώ τις ιδέες που υπέβαλες. Το ίδιο για τη δικαιοσύνη και τη μετάβαση σε... Θα ήθελα να σας πω το εξής για τον ειδικό εκπρόσωπο. Ε, όλο αυτό θα πρέπει να το δείτε, ε, το θέμα των ειδικών εκπροσώπων, ε, μέσα στα πλαίσια των όσων είπε η Φεντερίκα Μογκερίνη. Ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμένε κατευθύνσει προς κατεύθυνση που θέλουμε να συγκεκριμένες ιδέες ιδέες για την κατεύθυνση που πάμε. Έχουμε ερωτήσεις ε, και από τα κράτη-μέλη. Ε, ειδικό, ας πούμε, σύμβουλο για θέματα φύλου. Έχουμε το USR για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου όλα τα στοιχεία θα πρέπει να ενσωματώνονται εκεί, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλαδή. Αλλά αυτό το θέμα θα πρέπει να αποκτήσει, να μπει ψηλότερα, ας πούμε, στις προτεραιότητες μας, ε, σε όλες τις δράσεις της Ευρωπαϊκής υπηρεσίε εξωτερικής δράσης. Και πολιτικά θα πρέπει να είμαστε παρόντε όταν συζητώνται τέτοια θέματα. Για τη χρήση των ανεπάνδρωτων αεροπλάνων και ελικοπτέρων, τα drones. Ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η θέση των κρατών μελών. Υπάρχει μια μεγάλη προθυμία, για να το πω έτσι εφημιστικά, για να το συζητήσουν αυτό το θέμα σε, ευρωπαϊκές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ε, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, προσπαθήσαμε να το συζητήσουμε, αλλά δεν ήμασταν πολύ επιτυχείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ξεχνάμε. Για τα βασανιστήρια. Οι δράσει δεν είναι και πολύ φιλόδοξε. Και εγώ μάλιστα απογοητεύτηκα μετά από την, την ισχυρή από την κοινωνία των πολιτών όταν ήταν το χαρτί που μας έστειλαν, ήταν πάρα πολύ αόριστο και γενικό λόγο. Θα έπρεπε ίσως να καθίσουμε μαζί και να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο αυτό το έγγραφο. Για το χρονοδιάγραμμα. Λέτε ότι συχνά βάζουμε στο σχέδιο δράσης, ε, αναφέρουμε μάλλον ότι οι δράσεις αυτές είναι εν εξελίξη. Κοιτάξτε, οι προκλήσεις είναι τέτοιες που θα ήταν δύσκολο να πούμε ότι φέρει πίν στη δράση για την ενίσχυση των θεσμών για τα των εθνικών θεσμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το να θέσουμε μια προθεσμία όπως το 2017 ας πούμε είναι λίγο τεχνητό ας πούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες, ότι δεν υπάρχει υποβολή εκθέσεων. Ε, μου κάνει εντύπωση που είπατε ότι υπό το προηγούμενο σχέδιο δράσης δεν είχατε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για την πρόοδο που είχε επιτευχθεί να αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που αναφέρονται, αναφέρονταν σε εκείνο το σχέδιο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να αναφέρομαι τακτικά στην υποεπιτροπή. Το κάνουμε. Και προς την κοινωνία των πολιτών. Δεν θα πρέπει να κάνουμε κανένα αυτό το πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο εστιασμένα. Να εστιάζουμε, ας πούμε, σε συγκεκριμένα κεφάλαια του σχεδίου δράσης και να προσπαθήσουμε μαζί με την Κομισιόν να έρθουμε εδώ στο Κοινοβούλιο και να σας ενημερώνουμε. για τις, την εσωτερική και εξωτερική αξιοπιστία και την μετανάστευση. Αυτή η ιστορία, αυτό το θέμα βρίσκεται στον πυρήνα των συζητήσεων της Κομισιόν. Υπάρχει και μια ατζέντα για τη μετανάστευση που ετοιμάζουμε. Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος το ετοιμάζει με την βοήθεια της υπηρεσίας μας, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τομείς όπου μπορούμε να συνεργαστούμε πιο στενά. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την πρώτη παρατήρηση της κυρίας Λόχμπίλερ, είπατε ότι είναι πολύ πλήρες. Ε, νομίζω ότι ήταν και έπαινος και επίκριση ταυτόχρονα. Πολλοί ε, τομείς δεν έχουν ε, αναφερθεί για στρατηγικούς λόγους. Για παράδειγμα, δεν έχουμε θεματικά κεφάλαια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι καλύπτονται από άλλα κεφάλαια. Πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να δημιουργούμε έγγραφα για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά να επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην εφαρμογή. Γι' αυτό, για παράδειγμα, δεν καλύπτονται όλοι οι θεματικοί τομείς στο κεφάλαιο 2. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν αναφερόμαστε σε όλα τα είδη των διακρίσεων. Από την άλλη, θέλουμε να ε, έχουμε μία ε, συγκέντρωση των ε, προβλημάτων που αντιμετωπίζονται κάθε μέρα. Οι συνάδελφοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εργάζονται συγκεντρωμένα και με αίσθημα ευθύνη. Στο προηγούμενο σχέδιο δράσης, όταν είχαμε συγκεκριμένες δράσεις, χρονικά καθορισμένες, όταν είχαν ολοκληρωθεί τις ξεχνούσαν οι συνάδελφοι. Το να έχουμε λοιπόν συνεχόμενες δράσεις είναι ότι όλος ο κόσμος έχει το αίσθημα της οικειοποίησης. Όσον αφορά τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, είχαμε δύο συζητήσεις στην Home και το ίδιο ισχύει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα κράτη-μέλη θέλουν πολύ να ενισχύσουν τους τομείς αυτούς. Καλούμε όλους τους συμβαλωμένους να υποβάλουν συγκεκριμένες δράσεις, διότι είναι πολύ εύκολο να μιλάει κανείς για οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, είναι αρκετά δύσκολο όμως ε, να τα διασφαλίσει με στοχευμένες δράσεις. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο παρατηρήσεις να κάνω πριν να σας αποχαιρετήσουμε. Καταρχήν λείπουν κάποιοι συντονιστές και λείπουν και κάποια μέλη της ε, Επιτροπής μας. Ο κύριος Μπροκ, για παράδειγμα, με συγχωρείτε, ο κύριος Μπροκ, ε, θα το ε, εξηγήσω, ζήτησε να γίνει διευρυμένη συνάντηση του Προεδρείου της ΑΦΕΤ σήμερα το πρωί, την ίδια ώρα που συνεδριάζουμε εμείς. Κανονικά αυτό δεν θα έπρεπε να συμβεί, αλλά συνέβη και το Προεδρείο αυτό θα συζητήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, οπότε λυπάμαι πάρα πολύ που κάποιοι συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να έρθουν εδώ σε εμά γιατί είχαν αυτή την υποχρέωση και εγώ θα έπρεπε να είμαι εκεί αλλά προφανώς ε, η υποχρέωσή μου είναι να προεδρεύσω αυτή τη συνεδρίαση. Το δεύτερο, θα ήθελα επισήμως να ζητήσω συγγνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, γιατί δεν σας ζήτησα να καθίσετε εδώ στο Προεδρείο μαζί μας. Είστε και εσείς ε, ε, ένα κομμάτι του πάζλ και σχεδιάστηκε λάθος η σημερινή συνεδρίαση γιατί δεν σας καλέσαμε να κάτσετε εδώ δίπλα μας. Γι' αυτό και μόνο κατάλαβα ότι ενοχληθήκατε και δεν, μπορώ να, ε, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί εκείνη τη στιγμή αλλά το αισθάνθηκα, γι' αυτό ζήτησα από τη γραμματεία να σας πλησιάσει και να σας ρωτήσει. Εγώ δεν ήξερα καν ότι είχε τεθεί τέτοιο θέμα και ήξερα πως δεν είστε καν γραμμένοι στον ε, κατάλογο για να μιλήσετε. Τεράστιο το λάθος μας. Θα ήθελα να μας συγχωρέσετε και να σας πω πως καταρχήν θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο και πλούσιο το να είστε δίπλα μας, αλλά επίσης πως είναι κάτι το οποίο ήταν τελείως εκτός δικού μου πεδίου ελέγχου. Εν πάση περιπτώσει θα αναλάβω την ευθύνη και το συντομότερο δυνατόν θα προσπαθήσω να το λύσω. Εσείς πάντα είστε διαθέσιμος ε, και ειλικρινά είναι πραγματικά πολύ άσχημο αυτό που σας κάναμε σήμερα το πρωί. Εντάξει, έτσι το λέμε στα ισπανικά, ε, υπερβάλλω κάπως. Ε, πάντως λυπάμαι πάρα πολύ. Κύριε Γκοντζάτο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Ελπίζω το θέμα αυτό και το έγγραφό σας να το συζητήσουμε και πάλι μιλιά και θα μας καθοδηγήσει στις προσπάθειες που θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω πως ε, στην σύνταξη του εγγράφου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Υπηρεσίας Εξαιρετικής Δράσης θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πρόοδο. Θα σας καλέσουμε τότε και επιτέλους θα κάτσετε και εσείς δίπλα μας και ελπίζω θα είναι και συνάδελφοι εκτός αν τους ξανακαλέσει για κάτι ο κύριος Μπροκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Sí, Patrice, Oui, merci, σας ευχαριστώ για τα πολύ ευγενικά σας λόγια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε προσθέσει και πολλά, ούτως ή άλλως το βασικό θέμα είναι να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Ε, θα έχουμε πολλές ευκαιρίες λοιπόν να συνεισφέρουμε όπως συνεισφέραμε ούτως ή άλλως και στην εκπόνηση των εγγράφων για την Eh, mm. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, παρόλο που τελικά δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν πολλοί από τους σκιώδεις για την έκθεση της κυρίας Λοχπίλερ. Θα της δώσω λοιπόν απευθείας το λόγο για να μας κάνει μια παρουσίαση του σχεδίου αυτής της έκθεσης για το θέμα της ε, καταπολέμησης της ε, διακίνησης ανθρώπων στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Λοχπίλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να μοιραστώ μαζί σας ε, τις ε, πρώτες σκέψεις για τη δομή αλλά και για το περιεχόμενο του κειμένου. Έχουμε κάνει ήδη μια ακρόαση η οποία προσέφερε πολλά. Είχαμε και εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών, Διεθνών Οργανώσεων για τη Μετανάστευση, την κυρία Βασιλιάδου που είναι η συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα. Οπότε εξακολουθώ με την συλλογή ιδεών και καλώ όλους τους σκιώδεις να ε, συνεισφέρουν ε, όσο ακόμα επιθυμούν. Η έκθεση μιλά για τη μάχη, για την καταπολέμηση ε, της διακίνησης ε, ανθρώπων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογραμμίζω λοιπόν τρεις φορές πως μιλάμε για τα εξωτερικά σύνορα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε κοιτάξει σε βάθος ε, όταν συζητήσαμε την τελευταία φορά το θέμα της διακίνησης ανθρώπων. γιατί το επέλεξα, γιατί πιστεύω πως αυτή τη στιγμή το τράφικινγκ είναι από τις πιο κερδοφόρες και μεγαλύτερες εγκληματικές ε, βιομηχανίες παγκοσμίω. Ο ορισμός είναι εξής. Ορίζεται ως η προσέλκυση, μεταφορά, υποδοχή και εμπορία ανθρώπων ε, και η μεταφορά του ελέγχου επί των ανθρώπων αυτών με στόχο την εκμετάλλευση. ανεξάρτητα με αν το θύμα έχει συγκατατεθεί ή όχι και όταν το θύμα είναι παιδί τα αδικήματα αυτά είναι αυτομάτως κακουργήματα ε, τράφικινγκ όταν πρόκειται για παιδί. Είναι ένας πολύ στήρος τρόπος για να το περιγράψει κανείς, αλλά αν δει κανείς συνθήκες κατά τις οποίες, υπό ζουν αυτοί που είναι τα θύματα του τράφικινγκ είναι πραγματικά φρικτές. Είναι μια δουλεία. Στο παρελθόν στη ΣΥΠΑ λέγανε πως ο δούλος είναι μια επένδυση, έτσι. Έτσι τους θεωρούσαν ως μια επένδυση. Και αν κοιτάξουμε το τι γίνεται σήμερα, ε, μοιάζει να είναι ένα είδος δουλείας προς κατανάλωση. Και αν πεθάνουν οι δούλοι μας αυτοί και τι έγινε. Έχουμε έναν ε, παραδίπλα να χρησιμοποιήσουμε. Θεωρούν λοιπόν πως οι άνθρωποι είναι εμπορεύσιμα αγαθά και αυτό οδηγεί στις χειρότερες δυνατόν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάμε για θεμελιώδη παραβίαση της αξιοπρέπειας και της φυσικής και ηθικής ακαιρεότητας κάποιου ατόμου του δικαιώματος της, στη ζωή, στην ελευθερία και στην ασφάλεια για οποιοδήποτε άτομο. Ένας από τους στόχους της έκθεσής μας θα έπρεπε να είναι να ε, ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε η μάχη για την πάταξη του τράφικινγκ να αποτελέσει προτεραιότητα παγκοσμίω και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας έτσι ώστε να καταργήσουμε αυτή την απάνθρωπη πρακτική. Για την ίδια την έκθεση δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε χώρα η οποία να μην πλήττεται από το φαινόμενο αυτό. Άρα λοιπόν θέλουμε να ρίξουμε μια ματιά από την παγκόσμια οπτική γωνία για το τι είναι ακριβώ το τράφικινγκ, τι είδου κακοποίηση και εκμετάλλευση γεωγραφικά που τοποθετείται και ποιε είναι οι τάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στι τρίτε χώρες. Όταν είδατε το χρονοδιάγραμμα θα διαπιστώσατε πως είναι πραγματικά επίκαιρη η έκθεση αυτή γιατί έχουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την εξάλληψη του τράφικινγκ που λύγει το 2016. Ήδη λοιπόν αυτή τη στιγμή προετοιμάζουν την ε, νέα στρατηγική για τη μετά το 2016 εποχή. Οι συστάσεις από τη δική μας έκθεση θα μπορούν και αυτές να θεωρηθούν ως μια συνεισφορά στη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπογραμμίσουν πόσο σημαντική είναι και η πτυχή των εξωτερικών σχέσεων. Πώς έχω δομήσει την έκθεση. Καταρχήν, να δούμε ποιες είναι οι κυρίαρχες και οι ανανεώμενες τάσεις, τι γίνεται με το τράφικινγκ σε διάφορες περιοχές του κόσμου, Αφρική, Ασία, Λατινική, Αμερική, Μέση Ανατολή, ε, χώρες γειτονίας. Το δεύτερο στοιχείο θα μπορούσε να είναι τα οικονομικά στοιχεία για το τράφικινγκ, να δούμε την αλυσίδα ε, προσφοράς, ζήτηση, κατανάλωση, ξέπλυμα χρήματος, όπως επίσης και όλο το θέμα της ε, επιχειρηματικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, περιφερειακές εξελίξεις, κάποτε είναι πολύ ενδιαφέρουσες, στην ακρόαση μάθαμε πως υπάρχει μια σύμβαση για την περιοχή της ΑΣΕΑΝ, γιατί εκεί υποφέρουν πολύ κάποιες χώρες από το τράφικινγκ και έχουμε και κάποιες συστάσεις. Νομίζω πως χρειάζεται να κάνουμε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των εξή ε, σημείων. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει ένα κατάλογο χωρών προτεραιότητας επί του οποίου θα εργαστεί. Είναι ένα έγγραφο του 2009, έχουν ορίσει 10 χώρες ως χώρες προτεραιότητας και διαβάζοντας το έγγραφο λέει πως θα πρέπει να ελέγχεται σε τακτικά διαστήματα αν ο κατάλογος ισχύει ή αν θα πρέπει να έχουμε αλλαγές. Αυτό που βλέπω είναι πως δεν έχει γίνει τουλάχιστον σε τακτά χρονικά διαστήματα και διάβασα επίσης πως τα κριτήρια για το κατά πόσο μια χώρα είναι χώρα προτεραιότητας είναι, είναι το πόσοι οι πίκοοι της χώρας αυτής βρίσκονται μη καταγεγραμμένη στι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το Βιετνάμ, για παράδειγμα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί ε, Βιετναμέζοι χωρί ταξιδιωτικά έγγραφα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν ε, ε, η χώρα προτεραιότητα. Αλλά δεν μίλησαν για το τράφικινγκ που γίνεται με Βιετναμέζου προ την Κίνα ή άλλε χώρε τη Ασία. Άρα λοιπόν νομίζω τα κριτήρια θα πρέπει να συζητηθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά πολλά χρήματα στην μάχη για την καταπολέμηση του τράφικινγκ, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε πώς η χρηματοδότηση αυτή χρησιμοποιείται. Μήπως θα μπορούσε να είναι πιο στοχευμένη, μήπως θα μπορούσε να είναι πιο συνεκτική σε σχέση με άλλα ταμεία που διαθέτουμε και φτάνει όντως ε, εκεί που θα έπρεπε έτσι ώστε να προλαμβάνει τη θυματοποίηση ανθρώπων που πέφτουν στα δίχτυα των διακινητών. Μετά έχουμε το θέμα της επιχείρησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί έχουμε θέμα τράφικινγκ, και το λέω συσσαγωγικά τώρα, όταν βλέπει κανείς την αλυσίδα προσφοράς. Δηλαδή, επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται άτομα που είναι σήματα τράφικινγκ και να εξασφαλίσουμε πως έχουν πρόσβαση στην δικαιοσύνη, όπως επίσης και πως έχουν τα κατάλληλα ένδικα μέσα προσφυγής στα άτομα αυτά. Γιατί το λέω, γιατί η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θεωρεί πως τα θύματα βρίσκονται μόνο στο εσωτερικό μας. Όχι, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα θύματα και σε τρίτες χώρες και το τι του συμβαίνει ή τι δεν συμβαίνει. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα εξωτερικών σχέσεων. Μία προσέγγιση λοιπόν που στοχεύει κυρίως στα θύματα και όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τρίτα κράτη μπορούν να τα προστατεύσουν και να ευαισθητοποιήσουν τα ενδεχόμενα θύματα, να εντοπίσουν τις ανάγκες των θυμάτων και όλα αυτά είναι σημεία στα οποία χρειάζεται βελτίωση. Να δούμε και την πλευρά των κερδών, γιατί τα κέρδη που αποκομίζουν είναι τεράστια. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε τη διαδρομή του χρήματος και να δούμε τελικά ποιος κερδίζει έτσι ώστε με αποτελεσματικό τρόπο να πατάξουμε αυτό το έγκλημα. Στη γενική συζήτηση για τη μάχη κατά του τράφικινγκ θα πρέπει να δούμε και την πλευρά της ζήτησης. Και με ποιο τρόπο διώκουμε το έγκλημα αυτό. Δηλαδή, Europol, Eurojust, Frontex, αυτή είναι η θεσμή και οι οργανώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα. Για την αναφορά αυτή και για τη συγκεκριμένη έκθεση για τη διαδικασία. Η Επιτροπή Γυναικών μας είπαν πως θέλουν, υπο, πως θέλουν να συνδεθούν με την έκθεση αυτή υπό τον κανόνα του άρθρου 54. Είναι πολύ σωστό να ενδιαφέρεται η Επιτροπή ε, Γυναικών για το θέμα αυτό, γιατί θα πρέπει να εστιάσουμε και στο τι συμβαίνει με τις γυναίκες και τα κορίτσια Προτιμούσα όμως η Επιτροπή αυτή να το κάνει ως δική της γνωμοδότηση. Η Επιτροπή λοιπόν γυναικών θα υποβάλει μια δική της έκθεση όπου θα αναφερθούν στην εφαρμογή της ε, Οδηγίας 36 του 2011, όπου θα συζητήσουν και το θέμα του τράφικινγκ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι για την Επιτροπή Γυναικών αυτή είναι σωστή προσέγγιση, να μην κάνουν τη διάκριση δηλαδή, μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού. Ε, εμείς θα πρέπει να δούμε την πτυχή του εξωτερικού, γιατί είναι, είμαστε τμήμα αυτής της Επιτροπής και νομίζω το, πως αφού αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν μια γνωμοδότηση θα μπορούσαν να μιλήσουν και για τις δύο σελίδες που είναι η στρατηγική αυτής της οδικίας. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να διπλασιάσουν ε, τις προσπάθειές τους και να αντιγράψουν το όσα, τα όσα ήδη κάνουν σε μια νέα έκθεση. Για τα θύματα τώρα. Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι μόνο γυναίκες τα θύματα του τράφικινγκ δηλαδή καταναγκαστική εργασία. Εκεί η πλειοψηφία ε, των θυμάτων είναι αγόρια και άνδρες. Και ξέρω πως υπάρχει και μία έκθεση, με υπάρχει πρόθεση ε, η Προεδρία να γράψει στην Επιτροπή Γυναικών ε, λέγοντας ε, πως υπάρχει αυτό το θέμα, αλλιώς θα το δούμε στη διάσκεψη των Προέδρων. Έχουμε και, μία, και ένα αίτημα από τη Γραμματεία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, η οποία, επειδή κάναμε ακρόαση που ασχοληθήκαμε κυρίως με τα θύματα και δεν έγινε κατανοητό πως η δική μας ε, ακρόαση μίλησε για τα θύματα και τις εξωτερικές σχέσεις μας είπαν πως εφόσον πρόκειται για θύματα αυτόματα σημαίνει πως είναι εσωτερικό θέμα ελπίζω πως αυτή η παρανόηση από την γραμματεία της ΛΥΜΠΕ ε, να ξεκαθαριστεί θα ήταν καλύτερο εάν το επιθυμούν να συντάξουν και αυτή μια γνωμοδότηση αλλά δική μας έκθεση έχει να κάνει με θέματα εξωτερικών σχέσεων και δεν μπορούν να συνδεθούν μέσω του άρθρου 54. Έχω καταλάβει λοιπόν από τις όλες τις διαδικασίες πως εφόσον δεν έχει αποφασιστεί ε, το τι θα γίνει με το Άστρο 54 για τα συγκεκριμένα θέματα δεν μπορούμε να ετοιμάσουμε χρονοδιάγραμμα. Οπότε εγώ θα συνεχίσω με τα όσα κάνω στο περιεχόμενο και ελπίζω πως οι συνάδελφοι και οι υπόλοιπε ομάδες θα συνεισφέρουν καθόλου θα ήταν να τελειώσει φέτος, έτσι ώστε κάποιες από τις συστάσεις να ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την στρατηγική μετά το 2016. Ευχαριστούμε. Την κυρία Λοχμπίλερ, ποιο θέλει να κάνει κάποια παρέμβαση ή κάποια ερώτηση στην κυρία Λοχμπίλερ, ο κύριος Λίτς. Ευχαριστώ. από τον κύριο Άντι Κριστιαν, που είναι Ρουμάνος, ε, θα ήθελα να σας διαμηνήσω τις ιδέες του και τις σκέψεις του γι' αυτό. Η εμπορία ανθρώπων είναι σοβαρότατη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι αδίκημα κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οι προσπάθειες ε, καταπολέμησης ή μάλλον οι προσπάθειες ε, εμπορίας ανθρώπων έχουν εντατικοποιηθεί ε, και η προσπάθεια πολέμηση επίσης έχει εντατικοποιηθεί, αλλά είναι ανεπαρκής. Ε, τον εναρμόσουμε τα νομικά πρότυπα και να έχουμε πραγματική διεθνή συνεργασία για ποινικά θέματα είναι σημαντικό για να πετύχουμε σε αυτό το θέμα. Η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι ε, η, βασική πρακτική στην εμπορία ανθρώπων. Υπάρχουν όμως και ε, βίαιοι και καταναγκαστικοί γάμοι, χρήση ανθρώπων, ε, ε, σεξουαλική εκμετα... Ε, καταναγκαστική γάμη κτλ. Ε, συνήθως άνθρωποι από τις φτωχές περιοχές μεταφέρονται στις πλούσιες περιοχές. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς μέσω της οικονομικής και κοινωνικής ενίσχυσής τους. Μέτρα για τα ευπαθή άτομα του πληθυσμού, τα παιδιά, τις γυναίκες, τις εθνικές μειονότητες, τις μειονότητες, και του ετούντε άσυλο είναι πολύ σημαντικό. Η εκμετάλλευση τη εργασίας είναι όλο και μεγαλύτερη. Ε, θα πρέπει οι προσπάθειε καταπολέμησης ε, τη καταναγκαστική εργασία να είναι προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρχει προστασία και βοήθεια για να μην υπάρχει εκμετάλλευση όλων των ανθρώπων και των μεταναστών. Θα πρέπει η Κομισιόν να, μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας να χρηματοδοτεί προγράμματα ε, σε ξένες χώρες που όπου μπορούμε εκεί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ε, εμπορίες ανθρώπων. Να εστιάσουμε κυρίως στην προστασία και στη δίωξη σε διμερές επίπεδο θα πρέπει να υπογράφουμε συμφωνίες με τρίτες χώρες, ε, ρήτρε για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ε, εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και, της, ε, και του ευρύτατου στόχου καταπολέμησης οργανωμένου κλίματος. Θα πρέπει να έχουμε επίσης περιφερειακή συνεργασία για να καταπολεμήσουμε την εμπορία ανθρώπων, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια, στην χώρα της Ανατολικής Γειτονίας, στην ε, Λατινικές χώρες, στις χώρες Καρυδικής ε, και στην, ε, στις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ασίας. θα πρέπει να αφυπνίσουμε επίσης την κοινωνία μέσω της κοινωνίας των πολιτών που έχει σημαντικό ρόλο για να ανταποκριθεί σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η κοινωνία των πολιτών παίζει σημαντικό ρόλο γιατί εκθέτει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με την εμπορία ανθρώπων. Η αφύπνιση της κοινότητας, της διεθνούς, η υποστήριξη των θυμάτων, η υποστήριξη των κυβερνήσεων και άλλων, ε, το να διώξουμε τους ε, είναι πολύ σημαντικό. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι όχι μόνο πάροχοι υπηρεσιών, αλλά στρατηγική εταίρη στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή τέτοιων πολιτικών κατά της εμπορίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε καλή συνεργασία με την κυρία Λοχμπίλερ και με άλλους συναδέλφους για να υλοποιήσουμε τους ε, κοινούς μας στόχους που είναι η σύνταξη μιας καλής έκθεσης. Αυτά είπε ο συνάδελφος. Σας ευχαριστώ που θα τα λάβετε υπόψη σας και να σας τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, να συντάξουμε την έκθεση φέτος. Θα δώσω το λόγο στους επόμενους συναδέλφους για το πρόβλημα που έθεσε η κυρία Λόχ Μπίλερ για την Επιτροπή Γυναικών και την Επιτροπή Λίμπε. Πρόκειται να, για μια έκθεση που ασχολείται με άτομα που τα εμπορεύονται εκτό των σύνορων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι θέμα τη Ευρωπαϊκής Ένωση ειδικό, ούτε είναι θέμα ειδικό των γυναικών. Έτσι. Είναι γνωμοδότηση και των δύο επιτροπών, δεν έχει νόημα δεν ξέρω πώς θα το λύσουμε το θέμα, τελικά μια γνωμοδότηση τριών επιτροπών κτλ. Πάντω δεν την πρόεδρε που αποφασίσουν. Οι πολιτικές ομάδε. θα ζητήσω ότι από τη γραμματεία ή μάλλον οι γραμματείες των, των επιτροπών θα πρέπει να το συζητήσουν. Ποιο άλλο θέλει να πάρει το λόγο, εκτός από τον κύριο Οστεδίτσιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σκιώδηση συγγετριά μας Ρενάτε Βέπερ δυστυχώς παραβρίσκεται σε ψηφοφορία σε άλλη επιτροπή και γι' αυτό δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει εδώ τις θέσεις της. Εάν περιμένουμε λίγο μπορεί να φέρει κάποιες σημειώσεις. Θα ήθελα να πω όμως ότι εκτιμώ το καλό ξεκίνημα της Μπάρμπαρα και ελπίζω η έκθεση αυτή να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε αυτό, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια καλή έκθεση ε, με συμφωνία εισηγήτριας και σκιωδών εισηγητών. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Επειδή λαμβάνει σε μεγάλο βαθμό υπόψη την εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες. Και οι εν λόγω χώρες θα πρέπει να επιδείξουν βούληση και ικανότητα να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό όταν λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια. Και κάποιοι πόροι θα πρέπει να δεσμευτούν για ακριβώς αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ να δω τις ε, σημειώσεις ε, σύντομα της Ρενάτε, διότι και εγώ πρέπει να ψηφίσω, διότι είμαι αναπληρωτή στην Επιτροπή αυτή. Πάντως εκτιμώ τις προσπάθειες της Μπάρμπαρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σίγουρα μπορείτε να στείλετε και γραφτά τα σχόλιά σας. Κυρία Λόκμπιλερ, θέλει το λόγο. Ναι, και μετά θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της μυρίσιας διάταξης. Thank you. So there is not so much to add. Ναι, ευχαριστώ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Κύριε Λίντς. Νομίζω ότι οι παρατηρήσεις σας ταιριάζουν στην δομή της έκθεσης. Και επίσης αυτά που είπατε για την ε, εμπορία ανθρωπίνων οργάνων και άλλα θα είναι παραδείγματα που θα συμπεριληφθούν. Στην έκθεση συνδέονται πάντα όμως με, την εξ, ε, με τις εξωτερικές σχέσεις. Αυτά, ε, κύριε Οστρεβίτσιους, πάντως είναι αδύνατον να ολοκληρώσουμε την έκθεση για τις αρχές του καλοκαιριού. Στοχεύουμε μάλλον για ψήφιση της έκθεσης τον Νοέμβριο. Σας ευχαριστώ όλους. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης. Έχουμε μία ερώτηση της κυρίας Σαρτζεντίνη. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τον Ιτα Ιτζαμάρα από την Ζιμπάμπου Υπερασπιστή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος πήχθη στις 9 Μαρτίου, σχεδόν ε, πριν δύο μήνες δηλαδή, στο Χαράρε, την πρωτεύουσα της Ζιμπάμπουε. Ήταν ε, κεντρικός τέλεχος ε, της ε, ομάδας διαμαρτυρίας Occupy Africa και μετά την απαγωγή του δεν έχει ακουστεί τίποτα από αυτόν. Και εγώ και η οικογένειά του ανησυχούμε σοβαρά για την κατάστασή του. Τίθεται ακόμα το ερώτημα αν είναι ακόμα ζωντανός. Ερωτώ λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε για να ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση του Ιταϊζαμάρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα πιέσει την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε για να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαπιστώσει που βρίσκεται και να διασφαλίσει την απελευθέρωσή του και την προστασία της συζύγου του και πώς θα καλέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να προστατεύσει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσει την ελευθερία λόγου και συνεταιρίζεστε όλων των ανθρώπων, ιδιαίτερα υπό το φως της νέας ε, δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Νομίζω πως εδώ έχουμε εδώ και τον κύριο Καστίγιο, ο οποίος είναι επικεφαλής αντιπροσωπείας στην Ζιμπάμπουε. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά, αν μου το επιτρέψετε. Πρέπει να σας πω πως και εγώ συμμερίζομαι τις ανησυχίες που έχετε εκφράσει τώρα και ανησυχούμε πάρα πολύ για το πού βρίσκεται και για την ασφάλεια ε, του κυρίου Σαμάρα. Παρακολουθούμε την ε, κατάσταση στενά ε, εμείς στη Χαράρε και χρησιμοποιούμε κάθε ευκαιρία που έχουμε επί τόπου αλλά και στις Βρυξέλλες να είμαστε σε επαφή με την κυβέρνηση της Ζιμπάμπου για να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας και να υποβάλουμε έτοιμα οι αρχές να κάνουν ό,τι μπορούν έτσι ώστε να ανακτήσει την ελευθερία του. Είχαμε την ευκαιρία να δημοσιεύσουμε μια ανακοίνωση στις 11 Μαρτίου, δύο μέρες μετά που εγκρίθηκε. Είναι η αντίδραση, όπως ξέρετε, της κοινωνίας των πολιτών που έχει λειτουργήσει πολύ στο παρελθόν ε, και βοηθά την κατάσταση των όσων υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη να έχουν τέτοια δημόσια ε, στήριξη θα δημοσιεύσουμε και ένα ανακοινωθέν για να ε, γιορτάσουμε την ε, έλευση του πρώτου μήνα και μετά θα δώσουμε κάτι αντίστοιχο για τον δεύτερο μήνα. Ε, κάνουμε προσπάθειες και με τους ομολόγους μας στον Καναδά, στην Αυστραλία, με την κοινωνία των πολιτών και να σας πω πως σε σχέση με ε, προηγούμενες εγκρίσεις έχει αλλάξει η κατάστασή μας γιατί στο παρελθόν ξέραμε πού είχε χαθεί το άτομο, ε, τι του συμβαίνει. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία πληροφορία για το πού βρίσκεται ούτε καν οι υπηρεσίες ασφάλειας δεν έχουν κάτι να μας πούν. Αυτό που είναι θετικό είναι πως ο Αντιπρόεδρος διάβασε στις 11 Μαρτίου μία πολύ σκληρή δήλωση όπου είπε πως η απαγωγή αυτή είναι βαρβαρή, πράξη, πράξη βάρβαρη και πως η κυβέρνηση θα αναλάβει τις έρευνες ε, για την υπόθεση αυτή. Μία σφυριγγυλή δήλωση λοιπόν χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής και ελπίζουμε πως θα λυθεί το θέμα το με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και μπορεί να επιστρέψει ο κύριος Σαμάρ στην οικογένειά του. Thank you very much, Mr. Carro. I don't know if Madam Sargentini wants to add something or... Κυρία Σαργεντίνη, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Let me thank um, the Commission and the External Action Service for their... Να ευχαριστήσω την Κομισιόν και την ε, Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης για την απάντησή σας. Ε, πραγματικά εκτιμώ που είναι τόσο δραστήρια. Και ελπίζω πως η δράση σας εκεί και η δική σας δήλωση θα πιέσει την κυβέρνηση της Ζιμπάμπα. Σας παρακαλώ πολύ αν έχουμε καλά ή και κακά νέα να με ειδοποιήσετε αμέσω. Ευχαριστώ. Κάτι ακόμα. Δεν... Να περάσουμε λοιπόν στην ερώτηση κυρίας Λοκπίλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Μαλαισία. Καταρχάς, όσον αφορά την ελευθερία λόγου, θα ήθελα να ρωτήσω η Ευρωπαϊκή Ένωση τι δράσει έχει αναλάβει για να αποθαρρύνει την κυβέρνηση της Μαλαισίας ε, να παρεμποδίσει την ελευθερία έκφραση. Ο της Ε, είπε ότι θα ανακαλέσει την, ε, τον δρακόντιο νόμο του 1946 ε, και το 2014 επίσης είπε ότι όχι μόνο θα διατηρηθεί ο νόμος αυτός αλλά θα ενισχυθεί κιόλας. Πρόκειται για τον νόμο κατά της ανταρσίας. Γίνονται λοιπόν αυτέρετες έρευνες και έχουν απαγγελθεί καταγγελίες κατά 44 ε, ε, ατόμων ε, λόγω του ότι εξέφρασαν ελεύθερα την απόψή τους. Η 26η διάσκεψη κορυφής της ΑΣΕΑΝ πραγματοποιήθηκε στη Μαλαισία και η κυρία Μάλμστρομ ζήτησε γρήγορη πάυση της Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαλαισία. Και η Ευρωπαία... Η διαμεσολαβήτρια ο ε, Ράιλι ζήτησε μελέτη επιπτώσεων, ε, δεν θεωρήθηκε όμως ε, επαρκής για να καλύψει τι υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπονήσει εκθέσει για κάθε χώρα με την οποία έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πώς σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία σύναψης Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου για να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς μπορεί να εκπονηθεί ο δικό χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Μαλαισία, με τις αρχέ δηλαδή και με την κοινωνία των πολιτών πριν τη, στη σύναψη τη συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα εκπονήσει μελέτη αντικτύπου όσον αφορά τα δικαιώματα ε, στην Μαλαισία συγκεκριμένα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και οι Κομισιόν θέλουν να παρέμβουν. Ο Φράνκο Ολιβιερού, που είναι ο Front Desk Officer από τη Μαλισία και η κυρία Κόντσα από τη Γενική Διεύθυνση Trade θέλουν επίσης, θέλει επίσης να παρέμβει. Ε, μπορείτε να παρέμβετε με τη σειρά που προτιμάτε. Ε, είμαι ο επικεφαλής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μαλαισία ε, και μαζί με την συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου αποφασίσαμε να απαντήσουμε μισές-μισές ερωτήσεις. Εγώ θα μιλήσω για την ε, πράξη αυτή για την ελευθερία έκφρασης και η συναδελφός μου θα απαντήσει για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και το, τη συνιστόσα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την πράξη για την εξέγερση. Η ανταρσία. Μας ανησυχεί όλο και περισσότερο τα διαμοιβόμενα εδώ και 1,5 χρόνο από τα μέσα του 2014 με πάρα πολλές διώξεις, ε, κατηγορίες ε, που αφορούν πάρα πολλά άτομα. Αποφασίσαμε να αντιδράσουμε λοιπόν ε, διτά. Πρώτον, να εκδώσουμε μία δήλωση της ΥΠΑ της εκπροσώπου, θα επανέλθω στη δήλωση αυτή και αποφασίσαμε να στείλουμε και μηνύματα σε βαθμού αξιωματούχου κάθε φορά που έχουμε τη δυνατότητα σε διμερή ευκαιρία να συζητήσουμε με τους μαλέσιους ομολόγου μα για την δήλωση της είπα της εκπροσώπου. Εκδώσαμε δύο δηλώσεις, ε, μία ε, το Μάρτιο και μία τον Απρίλιο για την ε, πράξη αυτή για την εξέγερση και κυρίως για την ενίσχυση της πράξης που όταν τροποποιήθηκε στις 9 Απριλίου από το Κοινοβούλιο της Μαλαισίας. Ενδεχομένως έχετε δει αυτή τη δήλωση. Θα μπορούσα να τη διαβάσω πολύ σύντομα η Μαλαισία αποφάσισε να ενισχύσει την πράξη για την ανεργία αντί να την ανακαλέσει, ενώ είχε αναγγείλει ακριβώ αυτό, και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσει για την άσκηση τη ελευθερία έκφρασης, όπω αποδείχθηκε από το πώ εφαρμόστηκε η πράξη αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι φίλη της Μαλαισία, υπενθυμίζει ότι ο σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων είναι σημαντικά στοιχεία ενό δημοκρατικού συστήματο υποστηρίζουν την ανάπτυξη, ε, την ευμερία και την αρμονία. Αυτό το εκδώσαμε πριν από ένα μήνα, λιγότερο από ένα μήνα. Όταν η κόρη του αρχηγού της αντιπολίτευσης ε, ε, κρατήθηκε για μία νύχτα για ένα λόγο που έβγαλε στο κοινοβούλιο εκ μέρους του πατέρα της ε, και ίσως αυτό συνδέεται με την πράξη εξέγερσης, ποτέ δεν έχουν, έχουν διευκρινίσει οι αρχές, αλλά ήταν ένα παράδειγμα χρήσης αυτή της πράξης στο συγκεκριμένο άτομο. Το δεύτερο επίπεδο δράσεων είναι να στείλουμε μηνύματα σε ανώτατους αξιωματούχους, τον διευθυντή, ας πούμε, της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης όταν ο διευθυντή αυτός συζήτησε με, την, με τον Υφυπουργό ε, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων όταν ήρθε στι Βρυξέλλε πρόσφατα, θέσαμε το θέμα της ελευθερίας έκφραση και την ελευθερία λόγου. Και την αντίληψή μας ότι η χρήση και η ενίσχυση της πράξης ε, εξέγερσης ε, πηγαίνουν σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που θα επιθυμούσαμε. Υπάρχει ένας νέος πρέσβης της Μαλαισίας, της Βρυξέλλες και συναντηθήκαμε κατά επανάληψη, δηλαδή η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση μαζί του και του στείλαμε αυτά τα μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα ξέρω ότι έφτασαν στην Κουάλα Λουμπούρ μέσω του πρέσβη, τα ο πρέσβη. Από ό,τι καταλάβαμε με τις συζητήσει με τους συνομιλητέ μας είναι ότι ο βασικό σκοπό τη πρόσφατης τροποποίηση τη πράξη αυτή. Κατά την άποψή του ήταν για να εστιάσουν περισσότερο στην ε, φυλή και στην θρησκεία. Αυτό τονίζουν συνέχεια. Σε ό,τι αφορά ε, το Σαμπά και το Σαρουάχ, την, ε, τις περιοχές αυτές, το σημειώσαμε αυτό, ότι οι ποινές μπορούν να επιβληθούν με βάση ε, της, ε, την πράξη αυτή κατά της εξέγερση και μάλιστα μπορούν να είναι και πολύ ψηλότερε μετά την τροποποίηση. Αυτό είναι που μα απασχολεί πιο πολύ. Συνεργαζόμαστε σενά, με την Κουάλα ε, για το θέμα της Κουάλα μάλλον, και με χώρες οι οποίες πιστεύουν τα ίδια με μας για το θέμα της Κουάλα το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι οι Μαλέσοι συνομιλητές επιμένουν ότι με αυτή την τροποποίηση είναι σαφές ότι η πράξη αυτή για την εξέγερση δεν μπορεί να ε, εφαρμοστεί όταν υπάρχουν επικρίσεις ε, κατά της δικαιοσύνης ή κατά της κυβέρνησης, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν και υποτίθεται ότι αυτό είναι μεγάλη βελτίωση κατά την άποψή τους. Ευχαριστώ, Αγκολίβια. Καλημέρα σε όλους. Είμαι η κυρία Κόντσα. Είμαι ε, ε, του τμήματος που ασχολείται με την Νότια και Νοτιοανατολική Αφρική, Αυστραλία, ε, Ασία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Και θα απαντήσω στις ερωτήσεις για την ε, Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Για το δεύτερο στοιχείο της ερώτηση για τον οδικό χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα δώσω το, Λόγω, ξανά στον αδελφό μου την υπηρεσία εξωτερική δράση. Εγώ θα απαντήσω στο πρώτο και τρίτο ερώτημα. Καταρχά για το γενικό ερώτημα, για το πώ η Κομισιόν θέλει να χρησιμοποιήσει τη διαπραγματεύση για την ε, Συμφωνία Ελευθερίου Εμπορίου για να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στα ημαλαισία. Να ξεκινήσω γενικά υπενθυμίζοντα την ολιστική προσέγγιση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στι εξωτερικέ μα σχέσει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, θα πρέπει να καθορίσουν όλες τις ε, πτυχές τη δράσης, της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η εμπορική πολιτική είναι τμήμα αυτής της εικόνας που συμπεριλαμβάνει ειδικά, αλλά όχι αποκλειστικά, εξωτερική πολιτική και την αναπτυξιακή συνεργασία και τις εξωτερικές πτυχές των άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών. Η εστίασή μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες όχι μόνο προωθούν ε, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, αλλά βασίζονται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπνέονται από αυτό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για τι διαπραγματεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωση στη Μαλαισία, δεν ξεχνάμε ότι η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική κατευθύνεται για να προωθήσει το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο ε, στην παγκόσμια αγορά γιατί οι εμπορικέ συμφωνίε μπορούν σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία να συνεισφέρουν στη βελτίωση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες. Θεωρούμε ότι όταν έχουμε περισσότερο εμπόριο και εισόδημα έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και ότι η βιώσιμη ανάπτυξη σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε μακρόχρονες περιόδους, ε, μας οδηγεί σε βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεύτερον, με βάση την κοινή προσέγγιση για τη χρήση των πολιτικών ρητρών, η Συμφωνία τερικής Σχέσης και Συνεργασίας που διέπει τις συνολικές μας σχέσεις με τη Μαλαισία και που περιμένει όχι μόνο τη ρήτρα που αφορούν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι σημαντικό ουσιαστικό στοιχείο των σχέσεών μας με τη Μαλαισία, αλλά και μια ρήτρα μη εκτελέσεων, κατά των εκτελέσεων, που δίνει την ευκαιρία ε, μονομερώς να αναστείλουμε μερικός ή ολικώ τη συμφωνία αυτή. Ή οποιαδήποτε συμφωνία που συνδέεται με αυτή. Όταν οι διαπραγματεύσεις μας για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ξαναρχίσουν, εμείς θα πιέσουμε να συνδεθεί ε, η Συμφωνία εταιρική σχέση και η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Το λέω εάν και όταν. Γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή ε, δεν είναι εν εξελίξη με τη Μαλαισία, δεν είναι ενεργές, είναι ανενεργές. Και έχουμε έρθει σε επαφή ε, σε υψηλό επίπεδο με τη Μαλαισία για να δούμε αν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να ξαναρχίσουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το κάνουμε σε όλες τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Για τη Μαλαισία τώρα η Κομισιόν σκοπεύει να προωθήσει φιλόδοξες διατάξεις για να υπάρχει ε, διακυβέρνηση, ε, λογοδοσία και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, ούτως ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο που υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό αφορά και τους κανόνες για τη διαφάνεια και την άμεση εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή των διατάξεων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη που διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή με τη Μαλαισία. Θα ήθελα ξανά να τονίσω ότι η θέση της Κομισιόν είναι αυτή που σας είπα. Αλλά το θέμα είναι ότι οι διαπραγματεύσει με τη Μαλαισία είναι ανενεργές. Το αποτέλεσμα αυτό θα είναι αποτέλεσμα ε, διαπραγματεύσεων. Οι διατάξεις όμως για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι πάρα πολύ σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ε, συμπεριλαμβάνουμε σε όλες τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Θα περάσω σύντομα στο σημείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα τώρα και την μελέτη αντικτύπου. Και στο σημείο αυτό να κάνω μια γενική παρατήρηση. Κάναμε μια ανάλυση για το πώς ε, επηρεάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέτοιες μελέτες ε, χρησιμοποιούνται για να είμαστε σίγουροι πως η εμπορική πολιτική χρησιμοποιείται για να γίνονται σεβαστά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουν λοιπόν αναλυθεί επαρκώς τα ανθρώπινα δικαιώματα στην, στα πλαίσια όλων των εμπορικών διαπραγματεύσεων και λάβαμε εντολή να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μετά το 2011. Όμως, μία σκέτη αξιολόγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν συνάδει πλήρως με τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει για την καλύτερη νομοθεσία έτσι ώστε και ο αντίκτυπος στο περιβάλλον και στα κοινωνικά θέματα θα λαμβάνονται υπόψη με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις αξιολογίες και τις μελέτες που κάνει η Κομισιόν. Στο σχέδιο σύστασης που έκανε η Διαμεσολαβήτρια 26 Μαρτίου λάβαμε ιδιαίτερως υπόψη κάποιες ανησυχίες του καταγγέλλοντα και στο σχέδιο συστάσεως θα θα απαντήσουμε μέχρι τις 30 Ιουνίου στο θέμα που μας προώθησε η διαμεσολαβήτρια τώρα για το θέμα της Μαλαισίας. Και επειδή ακούστηκαν όλες αυτές οι ανησυχίες και λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων αυτής της διαπραγματευτικής ε, διαδρομής θα δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να καλύψουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποια είναι τα πιο σωστά εργαλεία όταν θα ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Θα κλείσω εκεί, θα δώσω το λόγο τώρα στον Φρανκ Ολιβίε για να μιλήσει για το θέμα του δικού χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τα επόμενα βήματα λοιπόν σχετικά με την ε, εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω καταρχήν πως αυτή τη στιγμή έχουμε μια συνοχιζόμενη στρατηγική για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, που ξεκίνησε το 2011 και ισχύει μέχρι το 2015. Σύντομα λοιπόν θα αναθεωρηθεί. Μάλλον το δεύτερο εξάμεινο του 2015 και στα πλαίσια της ε, σύνταξης μιας νέας στρατηγικής θα έχουμε και μια ε, διαβούλευση προκαταρκτική με την κοινωνία των πολιτών. Η αντιπροσωπεία μας στην Κουάλα Λουμπούρ αυτή τη στιγμή ξεκινήσει μια διαδικασία διαλόγου με τοπικές με καπαόμικρον για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα επαναλάβω όσα είπα για την νομοθεσία περί ανταρσίας. Θέλουμε να είναι ε, πολύ στενός ο διάλογος που έχουμε με τη μαλίσια στα θέματα αυτά. Ε, θέλουμε λοιπόν, επειδή η τελευταία προσπάθεια το 2011, να ξαναπεράσουμε σε συναντήσεις για το θέμα αυτό. Έχουμε ήδη ε, τοποθετήσει το θέμα αυτό στη συνάντηση των υψηλά στάμενων αξιωματούχων που θα γίνει με τη Μαλαισία τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες. Και ελπίζω πως εκεί θα ξαναξεκινήσει ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Νομίζω πάντως πως αν έχετε ερωτήσεις μπορούμε να απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις εξηγήσει. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να λάβει το λόγο. Πριν κλείσουμε. Όχι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Γεια σας. Για κάτι.